Welcome, friends. We'll start the meeting now. Καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Επισημένοντας ότι έχουμε να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες πλην της μαλτιζικής, Κροατικής και Κελτικής και αυτό σημαίνει ότι περνάμε στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Κοινή εξέταση τροπολογιών στις προτάσεις για αναθεώρηση των τριών εκ τριμερών υπηρεσιών. Ξεκινώντας λοιπόν με το Σεντεφόπ, δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Αν Σαντέρ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι στις 23 Αυγούστου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση νέου κανονισμού ιδρυτικού κανονισμού για την ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης, με διτό στόχο. Την εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων του υφισταμένου κανονισμού με μια κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και προσδιορισμό, επαναπροσδιορισμό των στόχων της υπηρεσίας αυτής. Θα ήθελα λοιπόν με τη σημερινή μου παρέμβαση πολύ γρήγορα να σκιαγραφίσω την εικόνα που δίνω αυτές οι 121 τροπολογίες που έχω λάβει για την πρόταση νέου κανονισμού. Δεν εντόπισα μεταξύ αυτών σημαντικούς φραγμούς ε, ή εμπόδια που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως ανυπέρβλητα. Συμφωνούμε όλοι μάλλον ότι είναι μάλλον ισορροπημένη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να ικανοποιήσει για την ικανότητα να προχωρήσουμε ε, μαζί παράλληλα για να ευοδοθεί το χέτερο δυνατό αυτή η έκθεση. Θέλω να αναφέρω επίση για τους σκιώδεις συγκητές ότι με χαρά σημειώνω τη δυνατότητα για συνεργασία και τη διάσταση για συνεργασία και επίση θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ε, συμμετοχή τους ε, στη δουλειά αυτή μέσω των τροπολογιών που κατέθεσαν. Εάν λοιπόν δούμε σε λεπτομέρεια τα σημεία των τροπολογιών, υπάρχουν διάφορα σημεία σύγκληση. Πρώτα απ' όλα τη σημασία στενή συνεργασία μεταξύ των τριών τριμερών υπηρεσιών με στόχο την αποτροπή των επικαλύψεων και την ενίσχυση των ε, συνεργατικών σχέσεων. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας ε, προσκαλείται ως, παρατη... προσκαλεί ε, παρατηρητή στη Eurofound, τη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ένα άλλο σημείο σύγκλησης έχει να κάνει με τους στόχους της υπηρεσίας, ενώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΔΕΦΟΠ την περιορίζει στο ρόλο μιας υπηρεσίας η οποία προσφέρει ε, τη συνδρομή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θελήσαμε στο αυτό επίπεδο να ε, δράσουμε το σύνολο των ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους ε, εθνικούς παράγοντες, κοινωνικούς εταίρους, κυβερνήσεις δηλαδή και βέβαια και εγώ αυτό ζητήθηκε μάλλον να συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσεις και σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Επίσης ο κοινό ρόλος του Συμβουλίου, του Διοικητικού και του Διευθυντικού ε, οργάνου. Σε αυτό συμφωνώ επίσης ε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σαν και ήριο ρόλο τον προσδιορισμό μιας στρατηγικής για την υπηρεσία ενώ ο διευθυντής έχει ως καθήκον την καθημερινή και διοικητική διαχείριση της υπηρεσίας. Άλλωστε είναι και αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικές με το προσωπικό της υπηρεσίας και ως εκ τούτου μπορεί να διορίσει αναπληρωτή διευθυντή. Επίσης ε, πολύ σωστά αγαπητοί συνάδελφοι οι υποβάλλοντες τροπολογίες σε σχέση με το θέμα των αρμοδιοτήτων που περνούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθυντή. Ένα άλλο σημείο συνένεσης έχει να κάνει με το ε, γραφείο επαφών, το σύνδεσμο της υπηρεσίας που συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ιδρυθεί στις Βρυξέλλες για να έχει τις επαφές η ΣΕΝΤΕΦΟΠ με τις άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως δεν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκαθιδρεί γραφεία σε διάφορα, να ιδρύει ε, γραφεία σε διάφορα πρωτεύουσε. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι αυτό της μετάφρασης. Ε, θέλουμε, εν γέννη δηλαδή, και πολύ το λένε με τις να εξασφαλίσουμε για την υπηρεσία της ΣΕΝΤΕΦΟΠ τη δυνατότητα να προσφεύγει ε, σε υπηρεσίες μεταφραστικές πέραν αυτών της μεταφραστικής υπηρεσίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχει μεγαλύτερη ευελιξία η ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Πολλά είναι τα σημεία λοιπόν που θα χρειαστεί να συζητήσουμε, πολλά είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να αναπτύσσονται περισσότερες αποκλήσεις, αλλά πάλι δυνατότητα και η διάθεση για συμβασμούς υπάρχει σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά αλλά και ανθρώπινα μέσα και ταυτόχρονα στη διάρθρωση του και τη αρμοδιότητα του Συμβουλίου του Διοικητικού. Επίσης θα ήθελα, Πρόεδρε, κλείνοντα να πω ότι να εκφρασώ την επιθυμία να μπορούμε να συνεργαστούμε με τους σκιώδεις ηγητές, τους αδέλφου ε, που έχουν ε, ε, τα θέματα της ΕΔΕΦΟΠ, αλλά και τους λοιπούς και οδησηγητές και συγκέντριες που έχουν αναλάβει τις άλλες υπηρεσίες. Γιατί η ιδέα μας ήταν να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για το σύνολο των υπηρεσιών. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι είμαι πάντα στη θέση σας, ότι είμαι πάντα πεπισμένη ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Thank you. Ευχαριστώ. αυτές, ε, αυτοί οι τρεις οργανισμοί θεωρητικά αποτελούν μέρος μιας κοινή συζήτηση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Από ό,τι κατάλαβα όμως, οι εισηγητές προτιμούν να εξεταστούν ξεχωριστά. Θα ήθελα να ξέρω αν συμφωνείτε. Θα συζητήσουμε τώρα λοιπόν για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, θα μιλήσουμε και για τους εισηγητές και μετά θα μιλήσουμε για, τα, για τους λοιπούς οργανισμούς. Λοιπόν, σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Πάβελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλω να σε ευχαριστήσω για τις κριτές γραμμές και την αρχική παρουσίαση. Χρειαζόμαστε να προσέξουμε να βασίζεται στο κοινωνικό διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να βρεθούν βιώσιμες λύσεις. Πρέπει να προσέξουμε όμως να μην το παρακάνουμε σε ό,τι αφορά το στόχο μας και με βάση τη χρηματοδότηση που υπάρχει. Ο ρόλος του ΣΕΝΤΕΦΟ πρέπει να εφαρμόσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και τις πολιτικές δεξιοτήτων και προσόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει ο οργανισμός να παράσχει τεχνογνωσία για τους πολιτικούς ηθήνοντες αλλά σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις κυβερνήσει και στους κοινωνικούς εταίρους. μείωση του προπολογισμού σημαίνει και μείωση της ποιότητας της δουλειάς του οργανισμού. Εμείς δεν μπορούμε λοιπόν παρά να συμφωνήσουμε με τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ε, ανεξάρτητη ε, εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί. Πρέπει να, ακολουθηθεί, να συνεχίσουν να υπάρχει η ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει βεβαίω να έχουμε πάρα κατά νου την υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Θα πρέπει να ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τον ε, τον διευθυντή. Βεβαίω ο διαχειριστή αυτός, ο διευθύνων σύμβουλο θα πρέπει ε, να ασχολείται μόνο με την καθημερινή διαχείριση. Συμφωνούμε επίση με την τροποποίηση ό,τι αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων. Για τι υπηρεσίε μετάφραση που απαιτώνται για τη λειτουργία του οργανισμού μπορεί να χρησιμοποιεί και εξωτερικού συνεργάτε για τι μεταφράσει του ΣΕΝΤΕΦΟΠ εφόσον ε, βεβαίω ε, έχουν υψηλέ προδιαγραφέ ε, και σε κοινωνικό επίπεδο και σε περιβαλλοντικό. Ελπίζω να συνεργαστούμε για το φάκελο αυτό και θα τα ξαναπούμε. Thank you. Ε, then I'll go ε, ε, Σας ευχαριστώ και κύριε Συντράτκα είναι η επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση του εγγράφου και για την σύνοψη που μας έκανε. Το πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε, ήταν πάρα πολύ καλό, καλά ισορροπημένο και η συνεργασία λοιπόν σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό ήταν ε, πολύ απλή. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε τώρα θα επικεντρωθούμε και επικεντρωθήκαμε στην ε, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και θα πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε άλλη επικάλυψη των δραστηριοτήτων. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι μία από τις, ε, ένας από τους οργανισμούς εκείνους που συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της επαγγελματική κατάρτισης και έτσι δίνει μία σημασία ιδιαίτερη στη διευκόλυνση έβρεσης απασχόλησης και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες του οργανισμού Αυτό θα πρέπει να στριχθούμε στις βέλτιστες πρακτικές του παρελθόντος, να βελτιώσουμε την εποπτεία, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγούσε στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Σοντεφόπ. Βρισκόμαστε σε φάση δημοσίων ακροάσεων σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς αυτούς, το Σοντεφόπ και τους άλλους οργανισμούς. Δεν έχουν επισήμως ε, βγει τα πορίσματα της διαδικασίας δημοσίων διαβουλεύσεων. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο προκειμένου να λάβουμε τα αποτελέσματα. Είμαι βέβαιη δε ότι τα πορίσματα αυτά θα μας ε, διαβεβαιώσουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ αλλά και η Πρόεδρος, η κυρία Χάρκιν δεν είναι εδώ βλέπω. Είναι κανείς που θέλει να πάρει Από την Μπα, δεν βλέπω κανέναν. Και έτσι λοιπόν, να πάμε στην QNGL. Η κυρία Κούνεβα δεν είναι παρούσα. Α, είναι. Συγγνώμη. Τώρα σας είδα, κυρία Κούνεβα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τις τροπολογίες που προσπαθώ να συμπληρώσω την πολύ καλή δουλειά της εισηγήτριας Κύρια Σάντερ, προσπαθώ να ξεκαθαρίσω ακόμη περισσότερο τη σημασία που έχει η λειτουργία του κέντρου χωρίς να υπάρχει επικάλυψη με τους άλλους συγγενείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνδικών Διαβίωσης και Εργασίας, το Eurofound και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκός για την Ασφάλεια και την Υγιεινή Συνεργασία. Και πιστεύω στην ε, προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Και ακριβώς επειδή η προσφορά του κέντρου στα ζητήματα της κατάρτισης είναι τόσο σημαντική, θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς και φυσικά στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και προτείνω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνεται και από το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου αλλά και να μετέχει πιο ενεργά στις αποφάσεις το Διοικητικού Συμβουλίου με έναν αντιπρόεδρο. Επιπλέον, η διαφάνεια των εργασιών του κέντρου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη αυτό και ζητώ την απομάκρυνση μέλων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αν διαπιστωτεί σύγκρουση συμφερόντων. Εφόσον η παροχή βοήθεια στα κράτη μπορεί να είναι κρίσιμη, δεν θα πρέπει να δίνεται μόνο σε επίπεδο εφαρμογή πολιτικών αλλά και σε προηγούμενα στάδια. Το κέντρο θα πρέπει να μπορεί να υλοποιεί και πιλωτικά προγράμματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης κενών στις πολιτικές μας. Έχω κατατέσει και μια σειρά τροπολογιών που επίσης βλέπω πως έχουν κατατεθεί και από άλλους συνάδελφους για τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων διορισμών από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και βεβαίως με λογοδοσία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλω στο κέντρο θα πρέπει να διαθέτει πάντα και τους κατάλληλους πόρους, υλικούς και ανθρωπιστικούς, για την ολοποίηση των που και στα πλαίσια της αποτελεσματικότητας αρκεί να διαθέσει γραφείο στις Βρυξέλλες αλλά και όχι σε άλλες πόλεις εκτός της έντρας του. Νομίζω ότι κινούμαστε σε αρκετούς, με αρκετούς συνάδελφους στην ίδια κατεύθυνση και τα έχουμε υπό την καταδίκηση της συγκήτριας ένα καλό αποτέλεσμα στο κείμενο που θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του κέντρου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που άργησα. Είμαι σκιώδης και για τις ε, τρεις ε, εκθέσεις και για τους τρεις οργανισμούς, άρα τα σχόλιά μου θα αναφερθούν και στους τρεις οργανισμούς είναι κοινή άλλωστε λίγο πολύ η προσέγγιση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιε ιδιαιτερότητε για κάποιου οργανισμού. Καταρχά. να σχολιάσω σε ό,τι αφορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για του οργανισμού. Να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Ακούσαμε ότι κοιτώντα τι διαθεσμικέ συμφωνίε για του οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την αρχή του προπολογισμού, τη δημοσιονομική αρχή και την αρχή ελέγχου για του οργανισμού και θα πρέπει να εκπροσωπείται και μάλλον το να εκπροσωπείται στο Συμβούλιο με οποιοδήποτε τρόπο ενδεχομένω να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων. Να το λάβουμε υπόψη αυτό. Αν το Κοινοβούλιο τώρα θέλουμε να έχει εμπειρογνώμονες, όπως γίνεται τώρα για παράδειγμα στον οργανισμό του Τωρινό, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά να είναι σαφής ο ρόλος τους. Να μην ανακύπτουν δηλαδή ερωτηματικά, γιατί υπήρχε και στο παρελθόν αυτή η αμφιβολία για το ποιο πληρώνει τι. Τώρα, γενικώ πώς για τους οργανισμούς. Θεωρούμε ότι στόχος τους θα πρέπει να είναι να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε κάνει λοιπόν και έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Έχουμε καταθέσει και τροπολογίες για την προστασία και τη βελτίωση ενδεχομένω τη ανεξαρτησία των οργανισμών αυτών. Και δημοσιονομικό πώ, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δουλειά του, την καθεαυτή δουλειά του. Έχουμε και κάποιε τροπολογίε επίση για την ισότητα των φύλων. ή σε εκπροσώπηση των φύλων στου οργανισμού αυτού. Να δούμε ενδεχομένω τη διατύπωση, να το θέσουμε κάπω πιο κομψά. Αυτό είναι όμως θέμα διατύπωσης, αλλά μας ενδιαφέρει η ουσία του θέματος. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η ισότητα της εκπροσώπησης των φίλων στην Επιτροπή, στο Συνέδριο και οπουδήποτε αλλού και στο δικό μας το θεσμικό όργανο. Επίσης, υποστηρίζουμε μέτρα που αποτελούν, αν θέλετε, την δομική βάση των συνεργασιών, των συνεργειών που θέλουμε να προωθήσουμε. Και εδώ έχουμε κάποιες τροπολογίες επίσης για το ρόλο του παρατηρητή. Υποστηρίζουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Επίσης, καταθέσαμε άλλες τροπολογίες για να διευκρινιστεί το θέμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πόσο συχνά ανανεώνονται, πόσο μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους. Αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν. Να δούμε και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και κάποιες μικρές τεχνικές τροπολογίες καταθέσαμε για την διαδικασία αναστολής. Μάλλον, συγγνώμη, παύσης ε, του ε, διευθυντή σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι τέτοιο. Είναι τεχνικές αυτές οι τροπολογίες για θέματα διαχείρισης, για θέματα ανεξαρτησίας, θέματα προϋπολογισμού. Εδώ καταθέσαμε λοιπόν ε, τροπολογίες για να υπάρχει ένας αναλογικός έλεγχος στα... στον προϋπολογισμό. Γιατί υπήρξε γενικώ ε, μια τάση να υπάρχει έλεγχος στους οργανισμούς, λες και είναι μεγάλη θεσμικά όργανα, με μεγάλους προπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλφαναλογικότητα. Δεν λέμε προφανώς ε, να τους αφήσουμε εντελώς ελεύθερους και να μην υπάρχει κανένας δημοσιονομικός έλεγχος, προφανώς και όχι. Αλλά θα πρέπει σε τελική ανάλυση η δουλειά τους να έχει να κάνει πιο πολύ με την καθεαυτή, το καθεαυτέο αντικείμενο τους και όχι τόσο πολύ με τα διοικητικά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Από το ΕΝΕΦ. Κύριε ο κύριος Μαρτέν την αντικαθιστά. Κύριε Μπιτζον δεν είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Χρησιμοποιήστε το άλλο μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό θέμα η αναδιαμόρφωση των τριών αυτών υπηρεσιών. Δεν καταθέσαμε όμως τροπολογίες και θα σας εξηγήσω το γιατί. Για να επαναλάβω αυτό που είχαμε εξηγήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, ε, άλλωστε παρατηρήσεις που βλέπουμε να συμμερίζονται όλοι οι βουλευτές. Πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες κάνουν πολύ καλές αναλύσεις, πολύ καλές εκθέσεις. Επαρελειμμένως όμως υπογραμμίζεται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητές τους. Όταν ε, πολλές φορές ε, ε, χαρακτηρίστηκαν αυτές οι υπηρεσίες ως κάτι που θυμίζει τους μεξικανικ... το μεξικανικό στρατό, δηλαδή πολυάριθμημένα αλλά χωρίς ε, λειτουργία, χωρίς δομή. Ε, και ενώ πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική κατάρτιση, συνθήκες εργασίας, συνθήκες υγιεινής, χωροεργασίας, παραμένουν εν τέλει οι ε, υπηρεσίες επικοινωνιακής δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρούμε, άλλωστε το έχουν επισημάνει και άλλοι, ότι από τις τρεις υπηρεσίες περισσεύουν οι δύο. Η μία δηλαδή θα αρκούσε να κάνει τη δουλειά αυτή κατά τρόπον αποτελεσματικό. Και με αυτή την παρατήρηση θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαντέρς για τη δουλειά της και να τη συγχαρώ γιατί με τις τοποθετήσεις της λέει εμέσως αλλά σαφώς ότι έχουν πολλά λατώματα αυτές οι υπηρεσίες στη δομή τους. Λοιπόν, δεν καταθέτουμε τροπολογίες, μεν παρακολουθούμε όμως μεγάλη προσοχή τις δικές σας και τις προτάσεις τους. Thank you. That means that Καλώς. Ρωτώ αν θέλει κανείς άλλος το λόγο, μόνο για το σαντιφόπο όμως, όχι για τις λοιπές υπηρεσίες. Άλλα σχόλια βλέπω δεν υπάρχουν. Κυρία Πάκουλα, Επιτροπή Γενική Διεθνή Απασχόλησης, έχετε κάτι. Κύριος, έχετε το λόγο, εσείς παρακαλώ. Δεν είναι η κυρία Πάκουλα, αλλά ο κύριος Μάς, ευχαριστώ πολύ. Ε, ορισμένα σχόλια μόνο. Κοινά βέβαια για τις τρεις υπηρεσίες. Ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε λοιπόν για τα θέματα ε, που επεσήμανε και η συγγήτρια. Θα εστιαστώ σε ορισμένα μόνο. Καταρχάς ο ρόλος της ε, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού σε σχέση με τη διαχείριση του προσωπικού. Υπόθηκε ήδη ότι οι προτάσεις αυτές προτείνουν ε, η διαχείριση ε, της καθημερινότητας στη δουλειά του προσωπικού να ανατεθεί στον διευθυντή. Αυτός νομίζω βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Αυτό το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση και αυτή η κοινή προσέγγιση είναι η δυνατότητα να ανακληθεί αυτή η εκχώρηση εξουσίας από το διευθυντή και νομίζω πολύ συμφωνώ με τις τροπολογίες του. Κύριε Λάμπερτς εξάλλου ε, μας το είπε ότι, είχε ότι προβλέπει και μια ιδιαίτερη διαδικασία. Αυτό ακριβώς πράττουμε λοιπόν και εμείς στην πρόταση της Επιτροπής. Δηλαδή προβλέπουμε μια διαδικασία δυνάμει της οποίας εάν διαπιστωθεί στην καθημερινή διαχείριση του προσωπικού, διοίκηση του προσωπικού του διευθυντή, το προσωπικό του, το, το επιτελείο του, να ανακληθεί αυτή η εξουσία και να περάσει και πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό άλλωστε ισχύει εν γέννη και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάθε νέα εκτελεστική ή αποκεντρωμένη υπηρεσία με τους κοινούς κανόνες όπως έχουν ανθεωρηθεί. Άρα θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες αυτό ως αρχή. Για την υπηρεσία μετάφρασης τώρα. Το μεταφραστικό κέντρο, σαν το θεσπίστηκε επί τούτου, δηλαδή προκειμένου να υπηρετεί τις ανάγκες για μετάφραση των υπηρεσιών αυτών. Έχει και τον αναγκαίο ποιοτικό έλεγχο και εάν εξωτερικευθούν αυτές οι υπηρεσίες μετάφρασης και υπονομεύεται το μεταφραστικό κέντρο και αυξάνεται το κόστος σε σχέση με το αποτέλεσμα, γιατί οι ίδιες αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα πρέπει να, επι, ε, ε, να επαληθεύουν ε, την ποιότητα του μεταφραζόμενου έργου και ως εκ τούτου θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σώμα. Α, συγγνώμη. Ενδεχομένως θέλει να προσθέσει κάτι η πριν περάσουμε στο επόμενο. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και να τους πω ότι τώρα με βάση τα διάφορα σχόλια θα προετοιμάσουμε ε, το τα συμβαστικά κείμενα. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους. Ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στο Eurofound το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαφύωση και εργασία, Ο κύριος Σομπόν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και του συναδέλφου λέει ο κύριος Τσαμπόν. Θα πρέπει καταρχήν να ευχαριστήσω όλου του σκιώδεις συζητητέ. καθώς και όσους ε, συνεργάστηκαν με τις τροπολογίες τους, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες, εξαιρετικά επικοδομητικές. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα, θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία, τον στρατηγικό προσανατολισμό, ε, την σχέση με τους πελάτες του οργανισμού αυτού που είναι και τα θεσμικά όργανα, τα κοινοβουλευτικά ε, αλλά και οι εθνικές αρχές αλλά και οι αρχές, ε, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν πραγματικά να βρουν πολλά χρήσιμα στοιχεία στο έργο της Eurofound. Εκεί συμφωνούμε. Η συνεργασία με τα άλλα τριμερή όργανα προφανώς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ καλό πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις τεχνικές πτυχές έρευνας ε, με διεθνείς πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως ο ΩΣΑ αλλά και άλλους. Και βεβαίως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Εγώ θα βελτιώσω το κείμενό μου χάρη στις προτάσεις σας. Τώρα κάποια μικρά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν ή κάποια ε, ζητήματα που χρήζουν συζήτησης. Παραδείγματο χάρη, το ζήτημα του υποδιευθύντη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πλειοψηφία που θεωρεί, όπως και εγώ, ότι ένας οργανισμός 100 ε, ε, εργαζομένων και βεβαίως ε, με τον περίπλοκο στόχο και καθήκον να εργάζονται για 450 εκατομμύρια ανθρώπους μπορεί λοιπόν κάλλιστα σε ένα τέτοιο οργανισμό να υπάρχει ένας υποδιευθυντής και πρέπει και να υπάρχει διότι μπορεί ο διευθυντής να χρειαστεί να απουσιάσει. Τώρα υπάρχει το θέμα των καθηκόντων του, υπάρχει το θέμα του ότι υπάγεται στο διευθυντή βεβαίω, ο υποδιευθυντή, και υπάρχει και το θέμα, του ορισμού του. Και εδώ πρέπει να, να είμαστε όσο γίνεται υπέρ της λειτουργικότητας ε, και του επαγγελματισμού. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ε, εγώ ήμουν υποψήφιος κάποια στιγμή για να αντικαταστήσω έναν υποδιευθυντή. Ο διευθυντής πέθανε και μετά ήταν να πάρω εγώ τη θέση του. Ήμουν υποψήφιος. Και τι δύο φορέ τελικά τη θέση την πήρε ε, ένας Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Για πολιτικού λόγου. Και υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι, πολύ καλύτεροι από μένα. Εν πάση το αποτέλεσμα είναι ότι ο διευθυντή και ο διευθυντή τελικά βρέθηκαν στα δικαστήρια, ο ένα κατά του άλλου. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε. Πρέπει να δείξουμε επαγγελματισμό και πρέπει να υπάρχει ένα επαγγελματικό σύστημα, αν θέλετε, ένα σύστημα με βάση επαγγελματικά κριτήρια για τον ορισμό του διευθυντή και του υποδιευθυντή. Τώρα, το γραφείο στις Βρυξέλλες, βεβαίως, σημαντικό να υπάρχει. Εντάξει, το Βερολίνο δεν είναι και τόσο μακριά. Γραφείο υπάρχει και λειτουργεί ήδη και από ό,τι κατάλαβα, ε, εμένα μου είναι εξαιρετικά χρήσιμο. από την προσωπική μου εμπειρία. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το να μπορεί δηλαδή το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί ε, αυτόν τον οργανισμό. Ε, Ω ποιο βαθμό όμως. Ο ίδιος ο πελάτης, το Κοινοβούλιο είναι ένα πελάτης, έτσι στην περίπτωση αυτή, να είναι στο Συμβούλιο και να συμμετέχει υπερβολικά υπερβολικά, σε υπερβολικό βαθμό στον στρατηγικό προσανατολισμό της, ε, του οργανισμού, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε βεβαίως τη χρυσή τομή. Είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί καλά, που είναι αξιόπιστος. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα ε, και βλέπω ότι στηρίζουν και άλλοι συνάδελφοι, είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υποχρησιμοποίησης της υποαξιοποίησης ε, αυτού του οργανισμού. Θα δούμε πώς θα το ε, εκφράσουμε αυτό, αλλά πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του Eurofound, να χρησιμοποιούμε το Eurofound γενικά πρωτού απευθυνθούμε σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες. Σίγουρα θα βρούμε ε, τη σωστή διατύπωση εδώ. Τι άλλο Τώρα υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εγώ δεν θέλω αυτό ε, να μας απασχολήσει υπερβολικά. Θα μπορούσε να έχει μόνο γυναίκες ο οργανισμός ε, και δεν θα ζητούσα ποσοστό ανδρών. Ε, το Κοινοβούλιο έχει κάποιες συμφωνίες για τις αντιπροεδρίες και βεβαίω θα μπορούσαμε να, να μπορούσε να ισχύσει το, το ίδιο και εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. πρόβλημα. Ε, δεν πρέπει, πάση η συζήτηση του πώ θα βελτιωθεί το Eurofound Found, να επικεντρωθεί στο πόσε άντρε και πόσοι άντρε και πόσε γυναίκε θα αποτελούν ε, τον οργανισμό αυτόν. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχουν δυσκολίε. Ένα άλλο σημείο τώρα, το οποίο βεβαίω δεν μπορεί να αποτελέσει σκόπελο στην προσπάθειά μα, αλλά το σημείο που υπάρχει απόκληση είναι αυτή η ιδέα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να έχει μια εθνική ε, προσέγγιση. Δηλαδή για τους 100 εργαζόμενους, 100 εργαζόμενους, οι 80 τόσοι να είναι από μια χώρα διότι πρέπει πάντα σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη στο Ειδικό Συμβούλιο. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει καν ευρωπαϊκή λογική. Θα μπορούσε να γίνεται αυτό ε, διαδοχικά ή ε, κυλιόμενα. Εφόσον θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θέλουμε περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θέλουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό δεν δημιουργεί μεγαλύτερο προπολογισμό προς τώρα χρήματα, είναι μια συνδυασία στον χρόνο. Αλλά γιατί, γιατί να, τι να το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συζητάμε γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Και θα συνεχίσω να εργάζομαι με βάση τις τροπολογίες και να συζητώ με όλους εσάς. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέντροβα δεν είναι εδώ, βλέπω. Την αντικαθιστά η κυρία Ριμπέιρο, όμως. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Την κυρία Σεντροβά εκπροσωπώ και άρα θα μιλήσω στα αγγλικά. Καλώς ορίζει λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δύο βασικούς στόχους, την ενημέρωση των στόχων των οργανισμών και μια κοινή προσέγγιση δεν θέλει να θίξει θέματα διαχείρισης και δομών διοίκησης ε, των οργανισμών, αλλά θέλει να διατηρηθεί αυτό το τριπλό, το τρίπτυχο σύστημα και να κρατηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μαζί με τους συστηγητές ε, του ΕΛΚ προτείνει τις εξής αλλαγές. Οι οργανισμοί δεν θα πρέπει μόνο να συνδράμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλους τους θεσμικούς ε, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και το Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλλον οι, δι, διευθυντές θα πρέπει να λαμβάνουν, να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις για τη διοίκηση και την ιστορική διαχείριση των ε, οργανισμών και θα πρέπει να ε, προσλαμβάνουν αυτό το προσωπικό. Και οι δύο ελεγκτές θα πρέπει να έχουν καθεστώς παρατηρητή και οι συντονιστές του κάθε της κάθε θα πρέπει να ενημερώνουν τα μέλη ε, για τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμών. Μπορεί να έχει μόνο ε, ένα γραφείο στις Βρυξέλλες και τέλος ε, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών μεταφραστικών υπηρεσιών. Αυτά ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Λόπες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια πρώτα. Εγώ συμφωνώ σε πολλά με τον εισηγητή και βεβαίως ε, να δούμε και ποια είναι τα σημεία ε, τριβής στις τροπολογίες. Οι τροπολογίες μας, της ομάδας μας δηλαδή, δίνουν κυρίως ε, έμφαση στην πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει το Eurofound, η τριμερής λειτουργία, στη διαχείριση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, κοινέ ε, σε πολλές ομάδες και με τον εισηγητή. Το βασικό σημείο απόκλησης ε, έχει να κάνει ίσως με τις τροπολογίες που σχετίζονται με, τον, με τη μείωση του αριθμού των εκπροσώπων στο Διευθυντικό Συμβούλιο του Eurofound. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μειωθεί ε, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να υπάρχει αυτό το επίπεδο αντιπροσωπευση των κρατών μελών στις εργασίες της Eurofound. Ο βασικός στόχος είναι να υπάρχει ένας διάβλος εργασίας κοινό, ένα διάβλος ενημέρωσης και χρήσης ε, του οργανισμού αυτού, όχι μόνο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκ μέρους των κρατών μελών. Ε, κανεί, κανένα από τα τρία μέρη, ούτε οι εθνικέ κυβερνήσει, ούτε οι επιχειρήσει, ούτε τα συνδικάτα δεν θέλουν αυτή τη μείωση. Ε, δεν νομίζουμε καν το Ευρωπαϊκό και το, το Ευρωπαϊκό Επιτροπή και το Συμβούλιο να το επιθυμούν. Εν πάση θα το συζητήσουμε. Ε, τώρα για τη μείωση του κόστου ε, σε σχέση με το θέμα αυτό. Κατά τη γνώμη μας αυτή η μείωση του κόστους δεν έρχεται να αντισταθμίσει ε, τις γνώσεις που θα χαθούν, τις γνώσεις ε, πολύ διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών πραγματικότητων ε, που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε σε πάρα πολλές τροπολογίες. Ε, μένουν κάποια σημεία να εξεταστούν. Υπάρχει το έργο της Eurofound, το οποίο πρέπει να στηρίξουμε η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, ο τριμερής χαρακτήρας ε, του οργανισμού, να ενισχυθεί το έργο και των τριών οργανισμών ε, μέσω του συντονισμού τους, ε, βεβαίως καλύτερο συντονισμό με διάλογους διεθνείς οργανισμούς, ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχει του απαραίτητου πόρου ο οργανισμό για να επιτελέσει το έργο του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εγγυηθούμε την εξαρτησία του, να αυξήσουμε τη, συμμετοχή στο Δυτικό Συμβούλιο ε, του Γενικού Διευθυντή, να ενισχυθεί γενικά ε, ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή στην καθημερινή διαχείριση του οργανισμού. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο. Δεν είναι εδώ ο κύριος Γερικέ. Ίσως κύριε Μάκεντερ θέλει να πάρει το λόγο στη θέση του. Όχι, κάνει λοιπόν από το ECR. Λίν Μπόιλεν. Από την ομάδα της Γκουα. Α, δεν υπάρχει εδώ κανείς από την ομάδα της ΓΟΕ. Η κυρία Λάμπερτ, λοιπόν, να πάρει το λόγο. Και είμαι σκιώδης Συγκεκριμένα και για τις τρεις εκθέσεις, γιατί θέλαμε μια έτσι συνεκτικότητα, μια ομοιογένεια. Για τα θέματα τα οποία ακούσαμε για το Δουβλίνο. σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του Συμβουλίου. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες και χαιρόμαστε που διατηρείται αυτός ο χαρακτήρας με πολλαπλά κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύουμε ότι αυτό είναι θετικό. Για να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις επιπρόσθετες, στα επιπρόσθετα γραφεία. Προφανώς, ε, υποστηρίζουμε το να υπάρχει ένα γραφείο στις Βρυξέλλες. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και ξέρουμε τι προστιθέμενη αξία έχει, αλλά δεν έχουμε καταθέσει τροπολογίες για να περιοριστούν, αυτό, να περιοριστούν τα γραφεία αυτά μόνο στις Βρυξέλλες. Αν υπάρχει λόγος να παρουσιαστούν επιχειρήματα για κάποια γραφεία αλλού, να τα ακούσουμε τα επιχειρήματα αυτά. Αυτά σε ό,τι αφορά τον οργανισμό του Δουβλίνου και θεωρούμε ότι τα σχόλια αυτά ισχύουν και γενικότερα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Γκέρικα. Όχι. Δεν έχετε κάτι να προσθέσετε. Η ευθυντή. Η κυρία Αγγιά. Ναι, ευχαριστώ, πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφα για την πρόταση της. Ε, η δουλειά μας θα πρέπει, αντιλαμβάνομαι, να εστιαστεί στη διατήρηση, και αυτό ήταν και ο στόχο μας, να εστιαστεί λοιπόν σε συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή περιορισμό του κόστους, ενίσχυση της διαφάνειας και εξορθολογισμό της λειτουργίας της υπηρεσίας και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και ο κοινωνικό διάλογος βέβαια αλλά και η ε, προαγωγή της απασχόλησης είναι κύριοι στόχοι. Έτσι λοιπόν συνεργάζεται και η Eurofound και ως εκ τούτου συνεργάζεται μαζί με τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ και την Ιώσα. Είναι πολύ σημαντικό να εξορθολογιστεί αυτή η δουλειά κατά τρόπον ώστε να μην κάνουν οι τρεις υπηρεσίε ε, το ίδιο πράγμα. Συνεργατικές σχέσεις λοιπόν, αποφυγή της επικάλυψης σε στόχους και δραστηριότητες, όχι μόνο μέσω αυτών των τριών υπηρεσιών, αλλά και έναντι της δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης σημειώνουμε ότι και άλλες ε, οργανώσεις, είτε εθνικού αλλά είτε διεθνούς χαρακτήρα, προσφέρουν αντίστοιχα αναλύσεις και δεδομένα για τις κοινωνικές, ε, πολιτικές και πολιτικές απασχόλησες. Όπως σε παραδείγματι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η ILO. Και έτσι πρέπει να εξασφαλιστεί μια δικτύωση μεταξύ αυτών των φορέων, ώστε η δουλειά τους να ενοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο χωρίς όμως να επικαλύπτεται η δουλειά της μίας με την άλλη. Ουσιώδου σημασία επίσης και άλλωστε το έχω περιλάβει στις τροπολογίες μου ε, είναι ο χρονισμός των δραστηριοτήτων της Eurofound ώστε να έρχονται οι προτάσεις της εγκαίρως και να είναι χρήσιμες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η, Ευρωπαϊκή, Eurofound να επιταχύνει τις δραστηριότητες της και να τις συντονίσει με αυτές τις ε, επιτροπές, όπως είπα, αλλά και των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πολλές φορές οι εκθέσεις δεν έρχονται πριν να οι εκθέσεις, οι μελέτες του Eurofound δεν έρχονται στα χέρια μας πριν να κλείσουν οι εκθέσεις δικές μας και άρα δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Το ίδιο για την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Είναι πολύ σημαντικό να τις έχουμε αυτές τις μελέτες εγκαίρως όπως άλλωστε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν την επικύρωση των ε, αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, και πρέπει να αποφευγεται η επικάλυψη εργασίας και πρέπει να γίνεται ε, πιο έγκαιρα η δουλειά και πρέπει να εξυγχρονιστούν τα μέσα μελετών και ερευνών, αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας και στη συγχρονή εποχή, με όλα τα μέσα, με το ίντερνετ, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τρόπο να υποφελεί για να βελτιωθούν οι μελέτες που ακόμη παραδοσιακό τρόπο διεξάγει η Eurofound. Τώρα θα ήθελα να περάσω στις προτάσεις που με μεγαλύτερη δυσκολία ε, θα βρεθεί λύση, πιστεύουμε, σε σχέση με τις άλλες εκθέσεις. Διότι εγώ έχω προτείνει οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων να περιοριστούν σε ένα μέγιστο εννέα μελών αντί να έχει κάθε κράτος το δικό του εκπρόσωπο. Και αυτό ισχύει και για τους εκπροσώπους οργανώσεων εργαζομένων που θα πρέπει να περιοριστούν με εναλλαγή αναδιετία, όπως γίνεται και στο, στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα και στον εκπρόσωπο της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγγνώμη. αντίστοιχα θα πρέπει να περιοριστούν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτοί οι εκπρόσωποι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο οι διορισμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν υπογραφής από τον ενδιαφερόμενο μιας δήλωσης περί συγκρόσεων συμφερόντων ε, σε σχέση με το καθήκον που αναλαμβάνουν προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Και από την εμπειρία που έχουμε τον κύριο Σαμπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, νομίζω ότι είναι εύλογο οι παρατηρήσει που έχουμε σε σχέση με ένα σύστημα και πρακτικές που πρέπει να αλλάξουν άρθιν. Από τέσσερα στα δύο χρόνια πρέπει να περιοριστεί η, η θητεία των μελών έτσι ώστε και να των μελών από τα κράτη-μέλη ε, και να υπάρχει αναλλαγή κάθε διετή έτσι ώστε να υπάρχει μια εναλλαγή και συμμετοχή ισόρροπη μεταξύ των κρατών μελών στη Eurofound. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μαρτάν. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα, γιατί αυτά που είπα νωρίτερα ισχύουν και για τις τρεις υπηρεσίες. Τελεία. Καλώς. Σχόλια. Μας. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπα προηγουμένως ε, για τον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή σε ό,τι αφορά την διαχείριση του προσωπικού αλλά και σε ό,τι αφορά το κέντρο μετάφρασης ε, αφορά και, τα, και τους τρεις οργανισμούς. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Επιτροπή, τους εισηγητές, τους και εισηγητές για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει για να υπάρξει μια ευθυγράμμιση των θέσεων επί των τριών προτάσεων. Όπως ελέγχθη νωρίτερα, έχει υποβάλει η Επιτροπή τις προτάσεις αυτές ως πακέτο, όχι μόνο της, ε, λόγω της φύσεως αυτών των οργανισμών, αλλά και διότι οι περισσότερες διατάξεις ε, αφορούν και, τις, και τους τρεις οργανισμούς και βεβαίως αυτό συνδέεται και με την κοινή προσέγγιση την οποία συμφωνήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2012. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να υπάρξει εδώ μια ευθυγράμμιση και στα τελικά κείμενα που θα συμφωνηθούν για τους τρεις αυτούς οργανισμούς. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα που ήθελα να θίξω έχει να κάνει με την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι η κοινή προσέγγιση προβλέπει όντως τη δυνατότητα, τη δυνατότητα αυτής της εκπροσώπησης όπου αυτό κρυφθεί σκόπιμο ε, να μπορεί να οριστεί ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο αυτό συνέβη παραδείγματο χάρη για κάποιες, κάποιους οργανισμούς ε, που χρηματοδοτώνται αποτέλει ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει μια αιτιολόγηση Γιατί δηλαδή να εκπροσωπείται κάποιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλει να προσθέσει κάτι ο συγητής. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίσω να εργάζομαι ε, με μεγάλη αισιοδοξία μετά από αυτά που άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν, βλέπω κοινά σημεία μεταξύ σας. Είναι το κοστούμι και η γραβάτα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα στην Ιγιου όσα. Παρακαλώ, ο εισηγητής έχει το λόγο. Ο κύριος Χόκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ως εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πολλά από τα ζητήματα που έθιξαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι καλύπτουν και την υπηρεσία αυτή συνεργαστήκαμε με τους κυρίους Σάντα Σαμπομπό και έχουμε πιστεύω μια κοινή προσέγγιση για τις τρεις αυτές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τους οργανισμούς, με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο καθένας τους βεβαίως. Ακολουθούμε λοιπόν μια τριμερή δομή που αντικατοπτρίζεται τόσο στους στόχους όσο και στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και συμφωνώ ότι αυτή η τριμερής δομή είναι όρος εκτρονού κόνευ για να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και για τα κράτη-μέλη και δι όλα τα κράτη-μέλη για τις εργασίες αυτών των οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν χρήσιμο έργο και μάλιστα ε, πρέπει αυτό το έργο να φτάνει σε όλους τους ε, εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το έργο αυτό. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τις σχέσεις με άλλες υπηρεσίες, Eurofund και Sendefop. Πρόκειται βεβαίω και για μέσα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και πρόκειται βεβαίως για την αντιμετώπιση των επικαλύψεων εργασίες, εργασίας. μεταξύ των οργανισμών. Όλα αυτά σαν κύριο μέλημα έχουν την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων που, προτείν, που προσφέρεται από τον Ευρωπαίο πολίτη στον προπολογισμό. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλουμε να κοιτάξουμε τα θέματα των στόχων του οργανισμού, των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής ε, ενημέρωσης, της σύγκρουσης των συμφερόντων και των ε, όρων σύνθεσης διοικητικού και εργασίας διοικητικού συμβουλίου και ε, διευθυντικών στελεχών. Προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία λοιπόν με όλους τους και όδης ηγητές, ε, τους ενισηγητές και πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε για να προσφέρουμε τις, μέγιστες, τις βέλτιστες δυνατές προδιαγραφές και το επίπεδο προστασίας στο χώρο εργασίας και της υγιεινής. Και ελπίζω ότι θα έχουμε έναν κανονισμό ευρωπαϊκό που θα συμβάλλει σε αυτό το στόχο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την κυρία Σάντερς, τον κύριο Σόμπο, για την πολύ συγκεκριμένη και επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους ε, σκιώδης ηγητές, όλους όσοι συνέβαλαν στη βελτίωση αυτής μου της εκθέσεως και ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Μπέκερ, μεταξύ των σκιωδών. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να εκφράσω ρητή ικανοποίηση για το ότι μπορέσαμε να συνδυάσουμε μια εξαιρετική δουλειά των τριών εισηγητών με πολύ υψηλό επίπεδο ομόνιας ε, και αντίστοιχο τρόπο εργασίας. Είμαστε σε ένα καθεστώς παρατηρητού. Έχουμε κάποιες βασικές ε, προτάσεις για τροποποίηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε προτάσεις ισοδύναμες από όλες τις ομάδες και αυτό είναι πολύ θετικό. Σημειώνω το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή ή της εκτελεστικής διευθύντρια στην περίπτωση της ε, όσα ε, και τις ευθύνες που πάντως δεν θα πρέπει να στερηθεί. Είναι απαραίτητο να έχουμε επαγγελματική ηγετική στελέχωση των οργανισμών αυτών για τη διαχείριση, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ισχύει αυτό όπως και για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Σημειώνω ότι αρκεί να έχουμε την υπηρεσία στις Βρυξέλλες, όχι ένα δίκτυο εκτεταμένο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, ε, ε, οι υπηρεσίες μετάφρασης που μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας από αυτούς τους οργανισμούς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι καθήκον αυτό ενός ε, ε, εκτελεστικού διευθυντή να το αποφασίσει, να το προσδιορίσει μια εκτελεστικής διευθύντριας. Επίσης η σχέση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προτάσεις που πιστεύω ότι θα μας οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους, όλους τους κοιόδης που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Ε, κύριε Κρίστενσεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έργο του έως τώρα. Όταν εξετάζουμε τις τροπολογίες ε, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ καλούς συμβασμούς για πολλά ζητήματα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η προστασία και η ενίσχυση του εταιρικού χαρακτήρα αυτού του οργανισμού θα πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της, τη σημαντική δουλειά της ε, αποτελεσματικά αυτός ο οργανισμός. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες τις οποίες ε, αναμένουμε να συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία των εισηγητών και των δύο τρεις για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για ζητήματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρενάτε Βέμπερ δεν είναι εδώ. Η κυρία Μπερμέιο, η Τζιν Λάμπερτ έφυγε. Δεν υπάρχει κανείς από το EFDD, μας το είχαν πει άλλωστε, και από το ENF ο κύριος Μαρτά επίσης δεν είναι εδώ. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν, έχουν, αν έχει σχόλια με βάση αυτά που άκουσε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το θέμα του κέντρου μετάφρασης νομίζω Ήδη εξήγησα γιατί υπάρχει αυτό το κέντρο και γιατί και από πλευρά τη ε, κόστος ωφέλεια είναι η καλύτερη λύση ε, για τον οργανισμό. Ε, θα ήθελα η τελευταία ευκαιρία που μου δίνεται για να, παρέμβω να τη χρησιμοποιήσω για να τονίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να σεβαστούμε την κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την, το θεσμικό διακανονισμό, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Ε, η καθημερινή διαχείριση προσωπικού είναι δουλειά του λογιστικού διευθυντή. Αυτό αναφέρεται σαφώς στην κοινή προσέγγιση, αποτυπώνεται και στις προτάσεις μας. Όμως, στις εξαιρετικές συνθήκες κατά τις οποίες αυτός ο εκκληστικός διευθυντής δεν θα μπορεί ε, να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να προβλεφθεί μία λύση ανάγκης και εκεί ακριβώς μπορεί ε, το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει πίσω αυτή την οξυδότηση προς τον Διευθυντή και να την αναθέσει σε κάποιο άλλο ανώτατο στέλεχος του προσωπικού. Είναι ένα σύστημα θεσμικό το οποίο έχει αποδείξει ε, την αποτελεσματικότητά του σε άλλα θεσμικά όργανα και γι' αυτό το επιλέξαμε στο πλαίσιο τη κοινή προσέγγιση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν αυτό δεν σημαίνει ότι ο διευθυντή ε, θα αλλάξει ε, τα καθήκοντά του ή θα αλλάξουν τα καθήκοντά του. Ο εκτελεστικό διευθυντή είναι αυτό που έχει την ευθύνη για την καθημερινή διαχείριση. Όμω για να μπορέσουμε να προβλέψουμε κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθηκοντά του διευθύντης, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα μπαίνουμε σε μια νομική διαδικασία, διότι δεν υπάρχει αυτή η λύση. Γι' αυτό ακριβώς ε, το συμπεριλάβαμε στην ε, γενική προσέγγιση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα η διαχειριστική ε, ή μάλλον το Γενικό Συμβούλιο να μπορεί να ε, αναθέσει αυτά τα καθήκοντα σε κάποιο άλλο ε, στέλεχος. Καλό λοιπόν τα μέλη να επαναξετάσουν πολύ προσεκτικά ε, το συγκεκριμένο στοιχείο, διότι όπως είπα είναι κάτι που θα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την κοινή προσέγγιση και άλλωστε είναι η πρακτική που ακολουθείται σε μια σειρά από οργανισμούς εκεί όπου έχουν μάλιστα ε, τροποποιηθεί ιστορική κανονισμοί για να προβλέπουν ακριβώ αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι που λειτουργεί πολύ καλά ε, επαναλαμβάνω πολύ σημαντική, σημαντικό το καθήκον του διευθυντή στην καθημερινή διαχείριση του προσωπικού. Ε, πολύ ωραία. Εξετάσαμε λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Η έγκριση της έκθεσης θα γινει 21-22 Ιουνίου. Να ευχαριστήσω την κυρία Σαντέρ, τον κύριο Τσαμπον και τον κύριο Χότς για τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν οι συγητές ε, έχουν κάποιο σχόλιο. Όχι. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της διάταξης Είμαστε και ένα τέταρτο μπροστά στο πρόγραμμά μας. Εγώ θα πρότεινα πάντως παρόλα αυτά να περάσουμε στο σημείο 6 πολιτικές περιελάχιστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας θα δώσω το λόγο στην κυρία Άγκια. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όδης εισηγητές και συναδέλφους που συνέβαλαν χάρη στις τροπολογίες τους στην συμπλήρωση αυτής της έκθεσης που είχαμε προβλέψει για τις πολιτικές ελάχιστο εισοδήματος με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας ο αριθμός των τροπολογιών που κατευθεί νομίζω αποτελεί και απόδειξη του ενδιαφέροντος ε, και της σημασίας που αποδίδεται όχι μόνο γιατί τα επίπεδα της φτώχειας στην Ευρώπη ενισχύονται εκθετικά και μάλιστα μας απομακρύνουν όλο και περισσότερο από την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020 που ήταν η μείωση της φτώχειας αλλά και γιατί ταυτόχρονα συνοδεύονται από το όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα της ανεργίας σε κάθε επίπεδο, φτώχεια των νέων, φτώχειας μακροχρόνιας και ταυτόχρονα από το απομάκρυνσης από τους στόχους της αυτοματοποίησης του 4.0 το επιπεδο 4 4-0 όπως το ονομάζουμε τέσσερις φάσεις και άρα εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της φτώχειας με στόχους απασχόληση όλο και περισσότερο και με όλο και αυξανόμενη σημασία. Προσπαθώ λοιπόν να αναλύσω και να κάνω προτάσεις συμβιβαστικές. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να σημειώσω απόλυτο θετική και επικοδομητική προσέγγιση από πλευράς των συναδέλφων, ε, την οποία διαπιστώνω, ως μια κοινή βούληση για την επίτευξη αυτών των σημαντικών στόχων, που είναι ακριβώς η καταπολέμηση της στόχης. Μπορεί να υπάρχουν βέβαια αποκλίνουσες θέσεις, προτάσεις διαφορετικές, που προκύπτουν από διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά πάντως έχουν σαν στόχο τον ίδιο ακριβώς, δηλαδή την καταπολέμηση της φτώχειας. Μαζί με τους συναδέλφους θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις διαφορές μεταξύ των θέσεών μας, ε, κάνοντας μια δουλειά στο δυνατόν πιο κοινή, πιο ενωμένη και απευθύνω έκκληση για την επίτευξη αυτού του στόχου που είναι κοινό στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Απασχόλησης, να κάνουμε δουλειά η οποία θα στέκει και θα αντιστέκεται απέναντι στα άλλα όργανα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πολλές φορές στο ρόλο αυτών της συναπόφασης που έχει ως ε, όργανο υφίσταται πιέσεις από πλευράς του Συμβουλίου και λιγότερο της Επιτροπής και πιστεύω ότι σε μια στιγμή κρίσιμη όπως αυτή την οποία ε, διανύει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο πιο ενωμένη στάση και θέσεις έχουμε ως Κοινοβούλιο, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τη συνεργασία και την υποχρέωση από πλευρά των λοιπόν θεσμικών οργάνων να λάβουν υπόψη τη δουλειά μας. Εμείς λοιπόν καλούμαστε τώρα να αποφασίσουμε εάν η δουλειά μας θα είναι μόνο μία ένδειξη, μία τοποθέτηση, η οποία όμως εξωτερώνει τόσο αυτός σκοπός και δεν αναπτύσσει περαιτέρω ε, συγκεκριμένες δράσεις ή εάν μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι το οποίο θα καταγράψουν ε, ως αποτέλεσμα η Επιτροπή και το Συμβούλιο σε μια πολιτική απασχόλησης για την Ευρώπη ως κάτι το οποίο θα προσφέρει περισσότερα από ότι ένα απλό έγγραφο κατευθύνσεων. Πρόκειται για μια δέσμευση, μια στράτευση ουσιώδη για μας ως ε, συνεισηγητών, ως κοινοβουλίου, μια στράτευση και μια δέσμευση που πρέπει να ε, λάβουμε, ένα ρόλο τον οποίο πρέπει να επιβεβαιώσουμε και αυτό το οποίο ζητώ εγώ από τα μέλη της Επιτροπής μας σήμερα είναι αυτό το έγγραφο το τόσο σημαντικό για αυτά τα πέντε χρόνια της ε, θητείας μας να οδηγήσει στην ανάπτυξη, σε δέσμευση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη μια νέα οδηγία, για να αποδείξουμε ότι δεν συζητούμε μόνο, γιατί βεβαίω έχουμε αποδείξει ότι με το να μιλούμε μόνο ένα αποτέλεσμα έχουμε μπορέσει να φέρουμε. Να αυξήσουμε τον αριθμό των φτωχών στην Ευρώπη. Πάνω από 120 εκατομμύρια είναι οι φτωχοί στην Ευρώπη, αυτοί οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πρέπει πλέον ε, και να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση αλλά και να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για κάτι το περισσότερο, για ένα εργαλείο συγκεκριμένο, ένα εργαλείο το οποίο θα στηρίξει αυτούς τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πια δεν μας ζητούν λόγια, αλλά συγκεκριμένες πράξεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στους Κιωδείς. Ο κύριος Μπαχ είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την κριτική της δουλειά και πιστεύω ότι πραγματικά και με τις συμβαστικές προτάσεις για τις τελογικές σκέψεις έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει ένα μεγάλο τμήμα της ε, δουλειάς. Η στρατηγική για το 2020, αν την κοιτάξουμε, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας και χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την ε, προστασία του κόσμου από τη φτώχεια και τον ορισμό της ε, φτώχειας της Eurostat. Συχνά τον επικρίνουμε τον ορισμό αυτό και υπάρχουν και κάποιες ε, τροπολογίες που έχουμε καταθέσει, αλλά είναι ουσιαστικά μοναδική ο μοναδικός ορισμός που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι στόχοι του της στρατηγικής το 2020 έχουν να κάνουν α, ακριβώς με την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης προφανώς είναι ο βέλτιστος τρόπος για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ενεργείας, αλλά και το ελάχιστος μισθός. Ο κατώτατος μισθός αποτελεί ε, ένα μέτρο δεδομένων των αριθμών των ανέργων. Αλλά οι κατώτατοι μισθοί έχουν να κάνουν και με την κοινωνική περίληψη έχουν να κάνουν και με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης κτλ. Κάποιοι ζητούν να είναι θεμελιώδης δικαίωμα αυτός ο κατατατός μισθός. Κάποιοι θέλουν αυτό να μείνει στην ε, διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αυτό το συζητάμε. Τα πιο πολλά κράτη έχουν κάποιες ρυθμίσεις για κατατατούς μισθού, αλλά με μεγάλες αποκλήσει προφανώς και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε με ποιο τρόπο μπορούν να βελτιωθούν τα ήδη υφιστάμενα συστήματα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι κυρίως το ευρωπαϊκό εξάμεινο και γι' αυτό καλωσορίζω το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την έκθεση του 2017 και για την κοινή έκθεση απασχόλησης που εγκρίθηκε τον Μάρτιο καλούν την εξασφάλιση, για την εξασφάλιση ότι τα κοινωνικά συστήματα θα δίνουν ε, σωστή υποστήριξη εισοδήματος. Και για να διαθέτονται πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες εξασφάλισης ε, μισθού και κοινωνικής ασφάλισης, η κυρία Αγκαία, ε, νομίζω ότι προτείνει στην έκθεση της όλα αυτά να ενισχυθούν μια έκθεση πρωτοβουλίας θεωρώ ότι δεν θα έχει κάποια σχηματική επίπτωση, δεν θα την λάβει υπόψη κανείς κάτι άλλο που είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Τα κοινά κριτήρια. Ποιος έχει πρόσβαση, τι εύρος εφαρμογής υπάρχει, ποιος εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση. Ε, τα κριτήρια ε, για να είναι κανείς δικαιούχος. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα με μειογένεια σε όλα τα κράτη ε, ένωσης. Κάτι άλλο που θα μας απασχολήσει είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Και εδώ ανακύπτουν μια σειρά από ερωτήματα. Πώς θα μπορούσε μια τέτοια οδηγία να διαμορφωθεί, τι παράγοντες, τι δείκτες θα περιλάμβανε, τι κριτήρια θα περιλάμβανε. Σίγουρα. Αυτό θα αποτελέσει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Νομίζω ότι συνολικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτό το ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να αποτελεί ε, ένα μέτρο για την απασχόληση και όχι να υποκαθιστά άλλες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπαχ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούτχερες Πυρετό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σημαντικά. Αύριο θα γίνει η προσυντηρία των σχεδόν συγκεκριτών βέβαια, αλλά υπάρχει ένα περιθώριο σαφώς για να υπάρξει συμφωνία για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση, διότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την εισηγήτρια, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και επίσης διότι τι περισσότερες πολιτικές ομάδες ε, συμφωνούν στα βασικά. Θέλουμε ένα νέο καθεστώς ε, κοινωνικής προστασίας ε, για αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους δεν αρκεί το παρόν πλαίσιο. Δηλαδή τα όποια επιδόματα ανεργίας. Σε αυτό το νέο λοιπόν σκηνικό όπου οι επιπτώσεις ε, από την ψηφιοποίηση παραδείγματος χάρη ή από άλλους ε, παράγοντες που οδηγούν στο κοινωνικό αποκλεισμό θα αυξάνονται. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας και να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ε, μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα ελάχιστο εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια για το ποιό θα έχει πρόσβαση σε αυτό το ελάχιστο εισόδημα. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση, να μην δημιουργούν δηλαδή ανυπέρβλητα εμπόδια, αλλά χρειάζονται κριτήρια. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Και εδώ πρέπει να βρούμε το κατάλληλο σημείο ισορροπίας. Ξέρουμε ότι είναι ε, μια έκθεση πρωτοβουλίας αυτή, δεν πρόκειται για νομοθεσία, αλλά πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να τροφοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδέες. Οι υπερβολικές ρυθμίσεις ή πολύ υψηλά προαπαιτούμενα ε, δημιουργούν ε, ε, μια αρνητική εντύπωση και μια απόρριψη. Από την άλλη βέβαια χρειάζεται, χρειάζονται τα όρια, χρειάζονται τα κριτήρια. Θα πρέπει αυτοί όμως που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το ελάχιστο εισόδημα να μπορούν ε, όσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές ε, να έχουν δικαίωμα σε αυτό το ελάχιστο εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν οι δημόσιες αρχές από τη στιγμή που προκύπτουν αυτές οι συνθήκες ε, κοινωνικού αποκλεισμού ή κίνδυνου κοινωνικού αποκλεισμού ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονται υποκειδομονία του ενδιαφερόμενου, ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για να έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο εισόδημα οι άνθρωποι αυτοί που το χρειάζονται. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να συζητήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι βεβαίω μια συζήτηση ουσίας, δεν θα το λύσουμε αυτό στην έκθεσή μας. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει απλά να γίνει μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει υποχρέωση τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν ε, μια τέτοια διάταξη και εκείνοι που πιστεύουν ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει μια υποστήριξη απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κοινωνικό προπολογισμό για αυτό το ελάχιστο εισόδημα. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας απλής σύστασης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνο, πυλώνα, μια ισχυρή κοινωνική διάσταση και ταυτόχρονα όταν μιλάμε για τις διάφορες μακροοικονομικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών να υπάρχουν και κάποια προαπαιτούμενα που θα πρέπει να πληρούν τα κράτη-μέλη σε κοινωνικό επίπεδο και είναι απαραίτητο να ορίσουμε τελικά ποιο είναι αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πρέπει να υπάρχει βεβαίω ένα σύστημα σεξουαλικό, δημόσιο, κατάλληλο, αλλά χρειαζόμαστε και αυτό το νέο ε, καθεστώς κοινωνική προστασίας το οποίο να αρκεί, να επαρκεί ε, για να εγγυηθεί ότι θα έχουν μια αποτελεσματική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτόν λοιπόν τον ορισμό θα πρέπει να παρέμβει ε, και ο κοινωνικό προπολογισμό. Τουλάχιστον μέσω των διαθροτικών ταμείων θα πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα όποια πλεονάσματα υπάρχουν ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ανοίγει η συζήτηση. Θα είναι δύσκολο να το κλείσει εδώ με αυτή την έκθεση, αλλά καλό ήταν να εκφραστεί η άποψή μας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Κέρικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, Λάουρα για τη δουλειά που έκανα. Νομίζω ότι κοιτώντα τι βέλτιστε πρακτικέ από όλα τα κρατη σίγουρα θα καταλήξουμε σε ένα σωστό, παρα... Ε, σωστό συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά ακούγονται ωραία και καλά. Εδώ στην Ευρώπη αγωνιζόμαστε για την κοινωνική ισότητα, για το ότι ο κόσμος πρέπει να έχει ε, ίσο και δίκαιο εισόδημα. Να σας υπενθυμίσω για το, τι είμαστε αρμόδιοι. Όσο και να με λυπεί αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στη Γερμανία ο μεγάλος συνασπισμός που εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, αν ε, θέλουμε δίκαιους ε, μισθούς, αυτό θα πρέπει να γίνεται στα εθνικά κοινοβούλια, στον Bundestag, όχι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εθνική αρμοδιότητα να ορίζονται αυτά τα πράγματα κατά το τιμιστή και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα, κοιτώντα στα 28 κράτη-μέλη, το τι γίνεται στην κάθε χώρα. Αν θέλουμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας, θα πρέπει να αγωνιστούμε στις πατρίδες μας ο καθένας. Στη Γερμανία έχουμε εργαλεία που ουσιαστικά εξωθούν κάποιες ομάδες του πληθυσμού στην φτώχεια, παρά που το γεγονός ότι υποτίθεται ότι ε, καταπολεμούν τη φτώχεια. Και αυτό προφανώς δίνει ε, επιχειρήματα στα ακραία κόμματα, στα ακροδεξιά κόμματα και σε τελική ανάλυση δεν αποτελεί καμία λύση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε ψευδοσυζητήσεις ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει να αποφασίσουν τα εθνικά κοινοβούλια και εκεί πρέπει να κρυθούν όλα. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι ε, στόχος μας να συγκεντρώσουμε τις βελτίστες πρακτικές. Και αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα διαθέσει ενδεχομένω στα κρατή-μέλη. Έχουν αλλάξει οι όροι εργασίε, αλλά αυτό θα πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο όπου υπάρχει η δικαιοδοσία. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν σε επίπεδο κρατών μελών. Το ελάχιστο μισθό, ο κατώτατο μισθό αποτελεί μια καλή ιδέα, αλλά προτού κατοχυρωθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιε είναι οι ομάδε ε, του κόσμου που επηρεάζονται. Γιατί οι ιδεολογίε δεν ε, οδηγούν ουσιαστικά σε σωστέ λύσει, αλλά σε νέε εξαρτήσει. Αυτό έχουμε να παρατηρήσουμε από την εμπειρία μα από τη Γερμανία. Δεν είναι μακροπρόθεσμες αυτές οι λύσεις πραγματικά για τις ε, ομάδες και του πληθυσμού που πληθούνται. Ουσιαστικά διαιωνίζονται οι εξαρτήσεις αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Τσαμπών έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Αγκαία όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για το θάρρος της, ε, για να που απασχολείται με ένα τόσο δύσκολο ζήτημα, ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Και το θάρρος της κυρίας Αγγεία είναι παράδειγμα προς για όλους. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία. Πολλά από αυτά που ελέγχθησαν πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα για να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Εγώ θα αναφερθώ στις τροπολογίες, μας και στην δική μας προσέγγιση ως ομάδα ALDE για το θέμα αυτό ε, της ε, του ελάχιστου εισοδήματο ω τρόπο καταπολέμησης της φτώχεια. Και στο τέλος θα αναφερθώ και στα σημεία διαφωνία. Το πρώτο που πιστεύουμε εμεί είναι ότι είναι εντελώ απαράδεκτο σε πλούσιες χώρες του πλανήτη όπως τα Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν αυτοί οι θύλακες φτώχειας. Αυτό δεν έχει ε, καμία νομιμοποίηση, καμία αιτιολόγηση ηθική. Όμως αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια για να βρούμε μια λύση. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο το ελάχιστο εισόδημα τελικά είναι χρήσιμο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχει τεθεί το ζήτημα. Αυτό συνεχίζει να τίθεται, διότι κάποιοι θεωρούν ότι πίσω από τα κονδύλια ε, που χρησιμοποιούνται ε, αυτό δεν αρκεί επασεπτώσει να ξοδέψουμε κάποια χρήματα και να με τη φτώχεια. Όπως ε, και με τον τρίτο κόσμο το ίδιο συμβαίνει. Κάποια χρήματα λοιπόν τα οποία διατίθενται, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά για να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η φτώχεια. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ηθική υποχρέωση, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα που μας λέει ότι ένα ε, εγγυημένο εισόδημα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εφόσον διαθωθεί σωστά, μπορεί πραγματικά να καταπολεμήσει την μεγάλη φτώχεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα τέτοιο ελάχιστο εισόδημα ένταξη, πείστε το όπω θέλετε, μπορεί όντω να καταπολεμήσει τη μεγάλη φτώχεια. Και αυτή είναι η πρώτη μας φιλοδοξία. Αυτό καταρχήν πρέπει να είναι καθολικό, έτσι. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για εργαζόμενους ε, και άνεργους, μιλάμε για νέους, μιλάμε για φοιτητές και βεβαίως μιλάμε και για συνταξιούχους. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο που θα διασφαλίζει την εκρίζωση αυτού που ονομάζουμε μεγάλη φτώχεια. Αυτή δηλαδή η οποία ουσιαστικά ε, βρίσκεται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι ήδη φιλόδοξο αυτό. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δύσκολα, περνάνε δύσκολα. Αυτό δεν πρόκειται να το λύσουμε όμως. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αλλά εδώ μιλάμε για επίπεδα φτώχειας μη αποδεκτά. Εκεί συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα, η φτώχεια σε σχέση με τα εισοδήματα είναι μόνο μία μορφή φτώχειας. Δεύτερον, το γεγονός ότι δίνουμε κάποια χρήματα δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Έχει κάποιο δυνατότητα να καταναλώσει κάποια ε, χρήματα, να τα διαθέσει και επίσης δίνει και μια αξιοπρέπεια. Λέει ότι τα χρήματα αυτά πλέον είναι δικά του και μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει. Τώρα, εκτός από την περίπτωση των συντάξεων, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι προσωρινά, όσο δηλαδή ε, υπάρχει αυτή η κατάσταση ε, ακραία φτώχειας, και με μια ενεργή πολιτική ένταξης. Συνοδευτική πολιτική ένταξης. Διότι θέλουμε να εντάξουμε το άτομο αυτό στην κοινωνία για να κρυζώσουμε τη μεγάλη φτώχεια. Το δεύτερο επίπεδο τώρα, και εδώ έρχεται η πρώτη δυσκολία, ίσως και η μεγαλύτερη. Εμείς θεωρούμε ότι ο ορισμός της φτώχειας και της μεγάλης φτώχειας κυρίως ε, σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον διαβίωσης του καθένα. Δεν είναι κάτι που να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, να μετρηθεί ε, σε μια ολόκληρη ήπειρο. Τώρα, υπήρξε μια ερμηνεία ατυχής αυτό του περίφημου 60%. Αυτό το 60% το να ορίσουμε έτσι τη φτώχεια οδηγεί σε παράλογα συμπεράσματα. Κάποιος που βρίσκεται λοιπόν κάτω από 60% του μέσου όρου ε, πάντα θα υπάρχουν φτωχοί εκεί, ακόμα και αν ε, τριπλασιάσουμε το μέσο μισθό. Δεν έχει νόημα αυτό. Όπως είπε και η Κομισιόν, ε, αυτό είναι ένα μέτρο διανομής, διανομής εισοδήματο. Δεν είναι κάτι όμως που μας βοηθάει να ορίσουμε τη φτώχεια. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε με απόλυτους όρους και όχι με σχετικούς όρους. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ε, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση και είναι βασικό ο άνθρωπος που βρίσκεται σε χρέα φτώχεια. Αυτό το νοικοκυριό, αυτός ο άνθρωπος, κατά πόσο έχει πρόσβαση σε βασικά ε, προϊόντα διατροφής, σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να καθοριστεί πολύ περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να δώσουμε εμεί έναν αριθμό εδώ δεν έχει νόημα. Αυτό λοιπόν το 60% είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει το κείμενο. Ε, επίσης οποιαδήποτε ποσοτικοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μας βοηθάει. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι δύο πράγματα. Να δημιουργήσει καταρχήν αυτό το δικαίωμα Μιλάμε για ένα εισόδημα, έτσι. Όχι για μισθό. Είμαστε σε μια πλούσια κοινωνία, μια κοινωνία ευμάριας. Έχουμε πολιτικές ε, φιλοδοξίες ως Ευρώπη, χρηματοοικονομικές. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να συνοδεύονται από αξιοπρέπεια. Αυτό όμως θα αποφασιστεί στο περιβάλλον του καθένα, στο πλαίσιο του καθένα. και η εφαρμογή προφανώς θα αφορά τα κράτη. Παραδείγματο χάρη, πολύ καλό το benchmarking, διότι όλοι έχουμε να μάθουμε από αυτό. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι διαφορετικέ καταστάσει σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να το απομονώσουμε, να πούμε Α, αυτό λειτουργεί πολύ καλά εδώ. Λειτουργεί καλύτερα σε ένα μέρο από ότι σε ένα άλλο. Ε, εξαρτάται όμω ε, ποιο είναι ο ο, εργατικο, ο εργασιακό ιστό, κατά πόσο υπάρχει βιομηχανία, κατά πόσο υπάρχει γεωργία κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι η υποχρέωση. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε βεβαίω και να συζητήσουμε. Ε, η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να δει ότι είναι επαρκές αυτό το εισόδημα. Ε, ότι μπορεί να εποπτεύει η Ευρώπη, να φροντίζει έτσι ώστε όντως αυτό το εισόδημα να καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Όμως ε, αυτό που έχει σημασία είναι κυρίως να τονιστεί το δικαίωμα, ότι είναι ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα με στόχο να τελειώνουμε με τη μεγάλη φτώχεια. Ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο. Και τώρα μιλάω ως Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν, έτσι. Ε, ενδεχομένως να μιλάω καν ως Άλντε. θα από την άποψή μου, δημοκρατικά. Εκεί όπου μπορεί να παρέμβει επίσης η Ευρώπη είναι στις οικονομικές ενισχύσεις. Διότι αυτά τα πράγματα συνδέονται. Δίνουμε δικαιώματα, δικαιώματα να πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να το απομονώσουμε αυτό. Δεν είναι όλες οι χώρες σε μια χρονική στιγμή όπου έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτά τα ελάχιστα σε όλους. Αυτό έχει να κάνει με την κινητικότητα, ε, βεβαίως η οποία δεν είναι πάντα θελούσια. Κάποιες χώρες μπορεί για μερικά χρόνια να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να είναι κάποια φυσική καταστροφή, μπορεί να είναι κάποια οικονομική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η ιδέα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μέσω των ταμείων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, όπως υπάρχουν αυτά τα ταμεία για το Fiscal Compact ε, ή για την άμυνα τώρα, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πετήσουμε και εδώ. Δηλαδή δημιουργούμε μια, δημιουργούμε μια Ευρώπη των πολιτών και υπάρχουν πολλοί συμπολίτε μας που δεν έχουν πιστεί για αυτήν. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αγορά. Και θα πρέπει να το μελετήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Προς αυτή την κατεύθυνση πάνε και τροπολογίες μου. Τώρα βεβαίω αν, αν δεν συμφωνήσει η ομάδα μου θα το λάβω υπόψη μου. Πάντως, πρώτον, να μιλήσουμε για αυτή την υποχρέωση, την ηθική, για το πώς θέλουμε να ζήσουμε στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε μεγάλη φτώχεια στην Ευρώπη. Να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν, ε, τι αποτελεί μεγάλη φτώχεια στην κάθε χώρα, ποιες είναι οι μεγάλες ανάγκες αυτό αποκλίνει από τη χώρα σε όλα για ιστορικού λόγους, κλιματολογικούς λόγου. και τρίτον να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτά τα ελάχιστα να μπορούν να καλυφθούν και οικονομικά με μία ακόμα κοινωνική ενίσχυση σαν και αυτέ που υπάρχουν ήδη. Το να προσπαθήσουμε πάντως να επιβάλλουμε ένα ποσοστό ή έναν αριθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτον δεν είναι εφικτό και επιπλέον θα υπάρξει πολύ σημαντική απόρριψη. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ πώς, να θα καταπολεμηθεί η φτώχεια στη Ρουμανία. Είναι μακριά για μένα. Δεν το ξέρω. Και οι Λατίνοι είμαστε βέβαια και οι δύο. Αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Δεν μπορώ να του πω εγώ, ξέρετε το 60% θα είναι το εισόδημα του μέσου μισθού. Μπορεί και με το 60% αυτό ε, η φτώχεια να μην αρκεί, να, να, μην καλύπτεται, να μην καλύπτονται τα, οι ανάγκες. Ή να υπερκαλύπτονται. Να το σκεφτείτε λοιπόν το θέμα αυτό. Ε, κατά τα λοιπά, καλό είναι να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση ε, για να φτάσουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν βλέπουμε κανέναν από την ΚΟΥ εδώ. Η κυρία Ντάνοκα, λοιπόν. Α, έχετε εκπρόσωπο από την ΚΟΕ. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ, καλημέρα και ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν σε άλλη συνεδρίαση, άλλη επιτροπή, εκπροσωπούσα τον κύριο Λόπες και θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν την άποψή του. Καταρχάς, κάτι που όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πολιτικής λιτότητας ε, που περιόρισε την δυνατότητα των κρατών μελών να δρούν στο κοινωνικό πλαίσιο και να επιτελούν τα κοινωνικά τους καθήκοντα παρέχοντας βοήθειας. Οι πολιτικές λοιπόν λιτότητας δεν ε, ήταν σωστή επένδυση και όλοι οι δείκτες ένδυας έχουν επιδεινωθεί, καθώς και η ανισότητα προφανώς. Η ανισότητα οικονομική και κοινωνική. Αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι πιο επίκαιρη ποτέ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Οι τροπολογίες που έχουν προταθεί για την ε, έκθεση εξασφάλιση συλλογική κοινωνική ευθύνη για την επιτόπιση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ε, το τι γίνεται με το κάθε άτομο ξεχωριστά. Θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια πολιτική για την απασχόληση και την ενοική περίληψη, συμπερίληψη συμπεριλαμβανομένων και μέτρων, μια σειρά μέτρων που θα εξασφαλίσουν τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων. Αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, δεν θα πέσει ο κόσμο ε, στην παγίδα τη ε, φτώχεια, στην παγίδα τη εξάρτηση. Μια κοινωνία με συμπερίληψη που θα εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οικονομικά δικαιώματα, τις συλλογικέ συμβάσεις, μια καθολική υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλεια, παιδεία χωρίς ε, δωρεάν παιδεία, ενίσχυση της ανάπτυξης για να αποφευθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Χρειαζόμαστε λοιπόν εθνικά τέτοια συστήματα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όποιος ε, Πλήρη τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες να μην υπάρχουν φλετικές διακρίσεις, διακρίσεις βάσει της ε, εθνότητας ή της ε, καταγωγής. Επίσης, θα πρέπει να βοηθούμε τον κόσμο σε φάσεις μετάβασης, όταν έχει βρεθεί δηλαδή σε μια φάση αποκλεισμού για να μπορέσει να επανέλθει στην ενεργή ζωή. Το μέσο εισόδημα το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τις πολιτικές κατά του μισθού για όλα τα κράτη-μέλη. 60% λοιπόν του μέσου μισθού θα πρέπει να είναι το όριο της φτώχειας για να εξασφαλίσουμε ότι τα εισοδήματα θα είναι πάνω από το όριο της φτώχειας. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία που καταπολεμούν τη φτώχεια θα έχουν μακροπρόθεσμες ε, ωφέλειες για την κοινωνία. Άρα δεν είναι αυτό επιβάρυνση, είναι επένδυση μακροπρόθεσμα για να υπάρχει κοινωνική περιληψή, ομοιογένεια και ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο Και τώρα να περάσουμε στην κυρία Ντάνοκα από του πράσινου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καταρχά θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, είναι μου προς την Λάουρα Τζέα και το θάρρος και την τόλμη που επέδειξε για να κάνει τις προτάσεις αυτές και για τη σημερινή συζήτηση. Και να συμφωνήσω με αυτά που ακούσαμε από τους φιλελεύθερους. Αυτό πιστεύω είναι το βασικό σημείο για τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην είναι κοινωνική ένωση όπως αναφέρεται στις συνθήκες. Πολλά γίνονται βασιζόμενοι στην αρχή του ανταγωνισμού. Αυτή του αμήλικτου ανταγωνισμού. Πιστεύω θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τις μεμονωμένες, ε, τα μεμονωμένα άτομα, τις οικογένειες ε, και τα κρατη Σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ε. Μεγάλο το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλούσιων. Βλέπουμε και τι γίνεται στο ιστορικό των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών. με την τελευταία διεύρυνση τα τελευταία 13 χρόνια από το 2004 διαπιστώνουμε ότι κλιμακώνονται, οξύνονται αυτές οι διαφορές, αυτό το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Μεγάλη εισρωή και των φτωχών ατόμων από κάποια κρατημέλη Προ άλλα κρατημέλη. Η δική μου χώρα έχει χάσει ένα τρίτο του πληθυσμού τη. Ήμασταν τρία εκατομμύρια, τώρα είμαστε δύο. Δεν ξέρω ποια είναι τα στοιχεία για τη Ρουμανία, μπορούμε να τα βρούμε, αλλά είμαι βέβαιη ότι είναι μεγάλα τα αριθμητικά ποσά και εκεί. Μεγάλα το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν φύγει και στην Πολωνία επίση. Έτσι έχει η κατάσταση. Και εκ παραλλήλου, η διαφορά μεταξύ φτωχών και πλουσίων, μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων, στη Λιθανία, στην ε, Ρουμανία, στην Πολωνία, είναι τεράστιο, τεράστιο το χάσμα. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής. Δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογίας, κύριε Τσαμπών. Είναι θέμα πολιτικής. Θα πρέπει να το επιλύσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό. Η δική μας λοιπόν θέση ποια είναι ότι θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες κοινέ αρχές. Κοινοί ορισμοί, κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Και όχι μόνο για το κατώτατο μισθό, το ελάχιστο εισόδημα, και αυτά ασφαλώς αποτελούν πρόβλημα, αλλά για το ελάχιστο εισόδημα το οποίο συζητάμε τώρα, θα πρέπει να οριστούν όλα αυτά τα ζητήματα και αυτή είναι η λογική της τροπολογίας που έχουμε καταθέσει για την παραγραφό 6. Δυστυχώς αυτό δεν περιληφθήκε έτσι στην αρχική μας πρόταση και έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την ε, τροπολογία. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί και έχουμε κάνει και μια σχετική τροπολογία είναι το ποιος θα είναι υπεύθυνο για όλα αυτά. Όχι μόνο οι πολίτες. Στο εντελογική σκέψη ε, όταν μιλούμε για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματο για του πολίτε. ξεχνούμε τους ε, λοιπούς κατοίκους, διαμένοντες στα κράτη-μέλη. Στη δική μου περίπτωση, στη Λετωνία, έχουμε 30% ε, του πληθυσμού που δεν είναι πολίτες, έχουν άλλο καθεστώς, δεν είναι πολίτες. Έχουν γενικά όμως δικαιώματα ίσα με αυτά των πολιτών της χώρας. Δεν θα μπορούμε να ξεχάσουμε τον κόσμο αυτό. Αυτό ισχύει και στην Εστονία. Έχουμε και κατοίκους ε, άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτός ο ορισμός. Θα πρέπει να μιλάμε για κατοίκους, πολίτες, διαμένοντες. Θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο σωστό. Και είμαι βέβαιη ότι στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση. Και το παλιό αυτό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα, του 2010, το οποίο μιλάει για το 60% τουλάχιστον 60% του μέσου εισοδήματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Να μην το ξεχάσουμε αυτό όταν θα καταθέσουμε καινούργιες προτάσεις για το ελάχιστο εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λίγη πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στον κύριο Μαρτά. Συγχαρητήρια, κύριε Μαλά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη εκ μέρου τη δόκτωρο Μελάν που βρίσκεται σε άλλη επιτροπή. Τελεία. Και έχετε κάτι να πείτε εκ μέρου τη. Όχι, καλώ ευχαριστώ. Και περνώ στου συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Ριμπέιρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς για τους συναδέλφους να πω ότι είμαι καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Σημειώνω ότι πολλοί είναι οι μαθητές για τους οποίους έχει ουσιώδη σημασία το ελάχιστο εισόδημα. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ακράδαντα ότι όλες οι οικογένειες, όλοι οι ιδιώτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν, πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα που θα τους εξασφαλίζει ε, μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό πάνω απ' όλα ισχύει για παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους. Και πρέπει ο μηχανισμός αυτός να αναπτυχθεί ως μηχανισμός ε, κοινωνικής ε, συμπερίληψης, αντιμετώπισης των αποκλεισμών, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Γιατί με όσα και να προσφερθούν δεν είναι δεδομένο ή να προταθούν, δεν είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν αυτές οι εγγύησεις ε, από τα κράτη για τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες πέραν των οικονομικών ε, που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας με υποστήριξη αυτής της εγγύησης. Αν δεν το κάνουμε αυτό, απλώς διαιωνίζουμε την εξάρτηση και το επίπεδο της φτώχειας. Το ελάχιστο εισόδημα λοιπόν πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να περάσουμε σε ένα μηχανισμό, πρέπει να μετατραπεί σε ένα μηχανισμό κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπερίληψης που δεν μπορεί απλώς να ε, αλλάζει όνομα, όπως είχαμε δει και στην Πορτογαλία. Χρειάζεται ένας πραγματικός μηχανισμός υποστήριξης για τους ανθρώπους που έχουν τόση ανάγκη. Ιδάλλως μόνο περισσότερη γραφειοκρατία δημιουργούμε. Ε, κυρία Ρεμπέρο, ευχαριστώ. Κύριος Φοντούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα και συγχαίρω τη συνάδελφα Ατζέα για την πρωτοβουλία της και την έκθεσή της. Καταρχάς θα ήθελα να αναρωτηθούμε ποιο είναι το όριο της φτώχειας χώρα. Γιατί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυτό θέλει να βοηθήσει. Να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει πείνα. Λοιπόν, άλλο είναι το όριο της φτώχειας στη Γερμανία, άλλο είναι το όριο της φτώχειας στη Γαλλία, άλλο στην Ιταλία και άλλο στην Ελλάδα. Γιατί παρόλο που έχουμε ενιαίο νόμισμα, δεν μπορεί ο πολίτης να αγοράσει τα ίδια αγαθά από τη μία χώρα στην άλλη. Όλοι λέμε ότι σε πολλές χώρες της Ένωσης εκατοντάδες χιλιάδες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό λοιπόν το όριο θα πρέπει να ξέρουμε για να δούμε και ποιο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν ένα ελάχιστο εισόδημα σαν μέτρο το οποίο θα είναι στην ουσία ένα βοήθημα γιατί για να μην πεθαίνουν οι πολίτες από την πείνα Ποιος όμως οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους στην εξαθλίωση και στη φτώχεια. Για μας είναι οι λάθος πολιτικές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι σίγουρα ο πρώτος παράγοντας, και δεύτερον τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Θα μιλήσω λίγο για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Η υψηλή φορολογία, οι περικοπές των κοινωνικών αγαθών, η τεκμαρτή φορολόγηση των πολιτών, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα, φορολογούνται επειδή είναι παντρεμένοι με 5.000, για 5.000 ευρώ. Επειδή την χάνει να έχουν ένα σπίτι για άλλες 3.800 ευρώ. Επειδή τυχαίνουν να έχουν και ένα σαραβαλάκι, ένα παλιό αυτοκίνητο δεκαετίας για άλλες 3.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικά άνθρωπος που δεν έχει εισόδημα ούτε ένα ευρώ φορολογείται για 12.000 ευρώ. Αυτή, αυτό το παράλογο δεν νομίζω να υπάρχει σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια έχει το, σκοπό του. Γιατί με αυτή τη φορολογία δημιουργεί η κυβέρνηση πλεονάσματα για την ικανοποίηση των δανειστών. Αυτά, αυτοί λοιπόν έχουν οδηγήσει στη φτωχοποίηση χιλιάδων Ελλήνων. Μόνο σε εθνικό επίπεδο και με άλλες πολιτικές μπορεί να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Καλή η έκθεση και σίγουρα θα αφυπνήσει κάποιους. Αλλά δεν περιμένω καμία σοβαρή πολιτική αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Are there other colleagues? Ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Μήπως η Επιτροπή. Έχετε να πείτε κάτι. Uh, no, no comment from the commission. Ουδέν σχόλιο. Καλώ ευχαριστώ κυρία Άουτζα, συγγήτρια. Ευχαριστώ για τα σχόλια των συναδέλφων και την υποστήριξη που εκφράστηκε. Ε, έχουμε νομίζω μια καλή βάση. Μου είπατε ότι, είμαι, ότι ήμουν θαραλέα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτοκτονικό αυτό που έκανα. Αν χαρακτηρίζεται δηλαδή από εσά ως αυτοκτονικό ή αν θεωρείτε ότι είναι κάτι το θετικό. Νομίζω ότι το θάρρο θα το δείξουμε με τη βούλησή μας να προωθήσουμε, να εισαγάγουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι η φτώχεια δεν αφορά ένα κράτος μέλος, είναι ευρωπαϊκή. 120 είναι τα εκατομμύρια των πολιτών που ζουν μέσα στη φτώχεια και αντιλαμβάνομαι μεν ε, τις ε, θέσεις ε, και τη λογική που σας καθοδηγεί, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινό πρόβλημα, αυτό συζητούμε σήμερα και πρέπει να ενωθούμε. Μπορεί να είμαστε κατακαιρματισμένοι στις θέσεις μας και τις πολιτικές μας σε κάθε τι άλλο, αλλά εδώ πρέπει ιδιαίτερα να επιμείνουμε να μείνουμε ενωμένοι. Χωρίς λοιπόν διάκριση γλώσσας, εθνικότητας, ε, πιστεύω θρησκευτικό ή άλλο, ή άλλο ε, πρέπει να δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα κοινό πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα είναι η φτώχεια. Και άρα η απάντηση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και σε αυτό πρέπει να αναλυφθούν κοινέ δράσεις. Για την παρατήρηση του συναδέλφου Σαμπούν. Βεβαίως έχουμε την κοινή αυτή θέση. Έχουμε ταυτόχρονα όμως και τη δυσκολία να δώσουμε ε, ένα μέσο όρο υπολογισμού αυτού του εισοδήματος. Ας αρχίσουμε λοιπόν να συζητούμε και να προσπαθούμε να αναπτύσσουμε κοινέ θέσει, συνθετικές προτάσεις. Αλλά πάνω από όλα εγώ λέω ότι έχει, έχει επισημανθεί ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της μεγάλη φτώχεια με δίκτες λοιπόν που μπορούν να καταγράφουν αυτή την ε, ε, κατάσταση. Θα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πιέτρο για όλη αυτή την υποστήριξη και βεβαίως συμφωνούμε πιστεύω σε πολλά. Με ικανοποίηση σημειώνω τα λόγια του συναδελφού Μπαχ, όπως και της κυρίας Ριμπέιρου, του κυρίου Ριμπέιρου, γιατί βλέπω ότι όσο και αν είμαστε πολλές φορές διχασμένοι στην Ευρώπη σε χίλιες διαφορετικέ θέσεις, σε αυτήν εδώ την υπόθεση προσπαθούμε από κοινού να βρούμε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ τη Τσανόκα. Ναι, Έχουμε κοινέ γραμμές πιστεύω και πάνω απ' όλα θα ζητήσω την υποστήριξή σας για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος έτσι ώστε να παρουσιάσουμε συνθετικές προτάσεις. Τόσο η δική μου η πατρίδα και η δική σας βλέπουμε σταδιακά να παρουσιάζουν μία ή μεταναστευτική Αμφίδρομοι, Έχουμε αφενός μεν πολλούς ε, μετανάστες που φτάνουν, ταυτόχρονα όμως ε, αδειάζουν οι πόλεις μας από τους νέους που φεύγουν. 10.000 είναι οι νέοι οι οποίοι έχουν αναζητήσει καλύτερες ε, ευκαιρίες σε χώρες άλλες. Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στην Ιταλία, όπως γνωρίζω βέβαια και την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ καλά, που επεσήμανε ο Σανερφος Φουντούλης. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα και εν τέλει εγώ θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ένα αποτέλεσμα κοινό για όλους. Λυπούμε. αν μου επιτρέπετε αυτή την παρατήρηση, που δεν ακούσαμε στο δύο λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που, κάνουμε αυτή την, ε, που κάναμε μια συνάντηση με την Επίτροπο Τάισεν, η οποία μας είχε ε, διαβεβαιώσει για μια θετική στάση που θα επεφύλασε στις προτάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Επερίμενα λοιπόν σήμερα έστω μια δειλή ένδειξη υποστήριξης, μια μετρημένη εκδήλωση υποστήριξης. Αλλά αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δείχνει πόσο πιο σημα... ακόμα περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένοι για να πείσουμε με ένα ισχυρό κείμενο, με ένα σαφές κείμενο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε, τις αρχές, το πώς η κάθε μια από τις πολιτικές ομάδες θέλει να τις προβάλλει βεβαίως, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι στους στόχους, στον ορισμό του τι σημαίνει να σώσουμε από το επίπεδο της φτώχειας αυτά τα 120 εκατομμύρια των φτωχών, έστω και αν ακούγεται κάπως κομική αυτή η έκφραση, πρέπει να δώσουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους αυτούς, στις γυναίκες, στα παιδιά, σε όλους τους φτωχούς και πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο το οποίο θα δείχνει ότι δεν έχουμε λησμονήσει το ρόλο μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να το λησμονήσουμε, πρέπει να στρατευτούμε έτσι ώστε να, κάνουμε ένα, να δώσουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και η Έχουμε ολοκληρώσει έτσι την πρωινή μας συνεδρίαση. Τρεις το απόγευμα τα ξαναλέμε. Τη παρουσία και της κυρίας Ηλιάνοβα από το ελεγκτικό συνέδριο για να συζητήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση ως προς το είναι αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της ανεργίας